ισχύει από το 18 Τετάρτου 18 και σύμφωνα με το, τη διάταξη 137 παράγραφος 2 του κανονισμού έχω αίτημα από ε, την ΦΑΜ σε σχέση με την ΟΚΕ για κάποια γνωμοδότηση όσον αφορά το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων και αν δεν έχουμε ενστάσεις τότε το αίτημα πρόκειται να